Άρχεται η συνεδρίαση. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αδελφοί, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, παρακαλώ ένα ερώτημα μονάχα σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, κύριε Πρόεδρε. Στις 12 είναι προσκεκλημένος ο Φίλιππος της Φουρβονίας για να λάβει